Έξοχα, έξοχα. Το σχέδιο ημερησίας διατάξεως λοιπόν ερμηνεύω τη σιωπή σα ω έγκριση, έγκριση των πρακτικών τη 7η Οκτωβρίου, εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Τώρα, έχω τη χαρά να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Σκοτίας, επικεφαλής είναι ο κύριος David Stewart. Σας καλωσορίζω και εσάς και τα μέλη. Είμαι λίγο, η φωνή μου είναι λίγο πραχνή Λοιπόν, David, σε ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω εδώ σήμερα. Και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω το λόγο στον David Stewart να μας ενημερώσει για αυτά που έχει να μας πει Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Στιούαρτ, που με καλέσατε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, καταρχάς, σας ευχαριστώ για την ε, εξαιρετική συνεργασία μαζί μας και θα ήθελα να σας καλέσω όλους και στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο για να παρακολουθήσετε και εσείς από κοντά όπως και εμείς σήμερα τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι για τη λειτουργία της Επιτροπής μας, όπως και για τη λειτουργία της δικής σας και για το έργο που έχετε κάνει στο Κοινοβούλιο. Πολλοί κόσμος, κυρία Πρόεδρε, αισθάνεται αποξενωμένος, απομονωμένος από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υπάρχει μια, ένα βάσιμο παράπονο για ανισότητα ε, και για το ότι οι αρμόδιοι φορείς και τα ιδρύματα δεν ακούν τη φωνή του, του κόσμου και τις απόψεις τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια έξοχη ιδέα να ξεκινήσουμε μια στενή συνεργασία στο πεδίο των αναφορών. Όλοι ε, σήμερα ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Ζουν για το σήμερα, προσπαθούν να βελτιώσουν το χτες και ευελπιστούν σε ένα καλύτερο αύριο. Τα τελευταία χρόνια ε, σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κοινωνικών δικτύων, του Facebook, του Google, αλλά είναι γνωστόν ότι η συμμετοχή στην πολιτική είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ έχουμε και επίση και χαμηλό ποσοστό συμμετοχή, αν και εμεί στη Σκωτία έχουμε 85% τουλάχιστον στο τελευταίο δημοψήφισμα που έγινε. Είναι πολύ ψηλό ποσοστό συμμετοχή. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικό μοντέλο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή Αναφορών. Εγώ θα ήθελα να ενισχυθεί πολύ περισσότερο η συμμετοχική διαδικασία στο θέμα των αναφορών. Ε, πολλές σε τοπικές αρχές και σε επίπεδο δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν επιτροπές και υποεπιτροπές αναφορών. Το κοινό το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει δώσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα, αλλά θα ήθελα είτε είναι στις Βρυξέλλες, το Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε στη Βαρκελόνη, είτε στην, ε, στο Λονδίνο να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και να ενισχύει ε, την λογοδοσία, την συμμετοχή και να ακούγεται η φωνή ε, των παραπώνων δεδομένου ότι οι πολίτες μας θέλουν τα κοινοβούλια τους να έχουν μία ε, άμεση επίπτωση στην πολιτική, στη στρατηγική των κυβερνήσεων τους. Η Επίτροπη μας δημιουργήθηκε το 1999 και συνεχίζει το έργο του προηγούμενου Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου του 1907, το οποίο βασιζόταν σε ένα πολύ παλαιότερο βέβαια του 13ου, 14ου αιώνα. Βεβαίω, όποιο θέλει να υποβάλει μία αναφορά, δεν πρέπει να υποβάλει μία αναφορά σε θέμα άσχετο το οποίο δεν μπορεί να χειριστεί και δεν είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, όπω έχουμε ζει τα τελευταία χρόνια, πολύ ενδιαφέρουσε αναφορέ. Παραδείγματο χάρη, αναφορέ που αφορούν την νομοθεσία της Σκοτίας, την ομολογία, ε, την προστασία θυμάτων από εγκληματικές πράξεις, προστασία των θυμάτων και ε, πολλές άλλες αναφορές οι οποίες διευρύνουν την ε, νομοθεσία του, της Σκοτής του Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου, της νομοθετικής εξουσίας καταβάλουμε μεγάλες προσπάσεις, να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, να, του, να τον ενημερώσουμε για την ορολογία, τη διατύπωση που πρέπει να ακολουθούν, για το πού, πότε και πώς μπορούν να επιβάλλουν την αναφορά και για το χρονοδιάγραμμα βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, προσωπικές διενέξεις ή εμπορικές ε, διαφορές, αυτές ανήκουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Προσπαθούμε επίσης να, να βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αναφορών, το οποίο λειτουργεί από το 2003. Σε αυτή την ψηφιακή εποχή ε, παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκολίες ε, στην υποβολή των αναφορών από πολίτες και Επίσης δίνεται η ευκαιρία μέσω του διαδικτύου να ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η κυβέρνηση του Ενμένου Βασιλείου έχει επίσης ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στο διαδίκτυο ηλεκτρονικών αναφορών και κάθε ε, αναφορά η οποία έχει πάνω από 100.000 υπογραφές πρέπει υποχρεωτικά να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, στο Westminster. Μία υπογραφή μόνο χρειάζεται για να εγκριθεί ε, μία ε, αναφορά. Δηλαδή όταν υποβληθεί για να φιλτραριστεί και να περάσει από την έγκριση χρειάζεται μόνο μία υπογραφή από τον αρμόδιο. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε που έχει υποβάλει μία βάσιμη ε, και λογική αναφορά έχει τη δυνατότητα να ακουστεί και να συζητηθεί. Είναι λοιπόν αυτή μια πλουραλιστική δυναμική, μια δυναμική πτυχή της πολιτικής. Πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή των αναφορών ε, ε, βοηθάει και ενισχύει τη δημοκρατία μέσα σε ένα εμπεδομένο δημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκε το κοινοβούλιο μας, έχουν έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση δραματικά. Έχουμε όλοι πλέον εμπειρία των κοινωνικών δικτύων, έχουμε όλοι τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones ή όσοι έχουν τέλος πάντων χρησιμοποιούν αυτή την προηγμένη τεχνολογία. Η οσοι εχουν τελο παντων έχει κάνει άλματα και από τότε που η Κομισιόν έχει ε, ε, διαμορφώσει τη νέα της ιστοσελίδα μπορούμε ε, να... Η Επιτροπή μας έχει ε, φτιάξει την ιστοσελίδα της, μπορούμε να διαχειριστούμε τις αναφορές ε, στο διαδίκτυο, online. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το σύστημα online, απευθυνόμαστε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, όχι μόνο στη Σκοτία, αλλά οπουδήποτε ζουν στον κόσμο. Είναι λοιπόν ευθύνη μας να διαμορφώσουμε και να παγιώσουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικών υποβολών και διευθέτησης αναφορών το οποίο να είναι προσβάσιμο και ευχριστό. Η μεγάλη πλειοψηφία η μεγάλη πλειοψηφία των ετούντων είναι, ε, προέρχονται από τη μεσαία τάξη και είναι άνω των 50 ετών. Υπάρχει λοιπόν ένα, ε, ένα συγκεκριμένο προφίλ ε, των ετούντων και των αυτών που του βάλουν αναφορές. Αυτό δείχνει ότι πάρα πολλά άλλα στρώματα του, των πολιτών μας είναι αποκλεισμένα. Εάν η διαδικασία υποβολής είναι περίπλοκη, αποθαρρύνονται οι πολίτες. Έχουμε και μία υπηρεσία υποστήριξη εμείς όσων των ενδιαφερομένων και είμαστε στη διάθεσή τους για κάθε ενημέρωση και βοήθεια. Στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινοβουλίου ε, ε, ε, ψηφίσαμε, συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμη η υπηρεσία αυτή. Έχουμε επίσης κάνει εκστρατείες και ε, ε, ημερίδες επιμόρφωσης στα σχολεία για να ενημερώσουμε ε, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευόμενους. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε κατά το βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις των πολιτών μας, να τους βοηθήσουμε στις αναφορές. Ξέρω ότι τα μέλη της Επιτροπή μας, ε, το μόνο, αυτό που τους ενδιαφέρει ολόψυχα είναι το συμφέρον των πολιτών, των Σκοτσέζων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ισότητα, την ε, δημοκρατική ε, συμμετοχή, να εισαγάγουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές, να εξασφαλίσουμε ισότητα μεταξύ των φύλων και όλες τις βασικές αρχές. Όπως σας είπα, ε, το θέμα των αναφορών ε, στις παλιότερες μορφές ε, κάποιου κοινοβουλίου είχε αρχίσει τον 14ο αιώνα. Από τότε έχει εξελιχθεί η ραγδαία και εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στους πολίτες μας έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην πολιτική διαδικασία βεβαίως ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις απαιτήσει τη σύγχρονη κοινωνία. Ποτέ δεν θα επαναπαυθούμε στις δάφνε μας σε ό,τι έχουμε επιτύχει και να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Συνέχεια εξελίσσεται και η τεχνολογία και οι απαιτήσει και οι ανάγκες. Πιστεύω ότι σας έδωσα μία ιδέα του, του έργου μας, του τι κάνουμε, των στόχων μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Mr. Stewart for Σας ευχαριστώ κύριε Στιώτ για μια πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση των εργασιών της Επιτροπής σας και είναι εντυπωσιακό το ότι διαρκεί αυτό από τον 14ο αιώνα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από σας και ακριβώς ε, γι' αυτό είσαστε εδώ. Προσπαθούμε να μάθουμε από το τι συμβαίνει στα κοινοβούλια των κρατών μελών και σε μας για τις αναφορές. Νομίζω ότι το τεχνικό σημείο έχει ρυθμιστεί. Για να ακούτε πρέπει να φορέσετε τα ακουστικά.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 Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά ο μισθός του staff in the petitions committee and the advice and guidance that they can give to petitioners really helps the system and helps the process. Είναι ο διπλός από τον μισθό που παίρνουν οι δικοί σας άσως προφανώς. Mrs. Curtin Darling. Thank you very much and Σας ευχαριστώ. Η κυρία Darling. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις Επιτροπές Αναφορών άλλων κοινοβουλίων και να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, πράγματι θα ήθελα να σας επισκεφθούμε, να δούμε πώς τα καταφέρνετε. Είναι μία ώρα από εκεί που μένω εγώ και θα έρθω με μεγάλη ευχαρίστηση. Ε, πολλοί από τους αναφέροντες, τους οποίους ε, εμεί αντιμετωπίζουμε και θα δείτε και εσείς στην επίσκεψή σας, είναι πολλές φορές ε, άνθρωποι μετανάστες εγκατεστημένοι σε άλλες χώρες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ε, τις οποίες δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς δέχεστε αναφορές από κατοίκους άλλων, από, ε, από πολίτες άλλων χωρών που κατοικούν στη Σκωτία να πω ότι ανεξαρτήτως από που ζεις μπορείς να αναφερθείς στο κοινοβούλιο μας εφόσον έχει κάποια σχέση με τις δράσεις ε, της ε, κυβέρνησης της Σκοτίας ή ε, γενικότερα της πολιτικής γύρω από τη Σκοτία και την υπόλοιπη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εμείς να πούμε ότι εκπροσωπούμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και πολλοί που ζουν σε άλλες χώρες ενδιαφέρονται με αυτά τα οποία κάνουμε. Έχει σημασία να έχουμε ένα δίκτυο κοσμοπολίτικο, διεθνές και να επαναλάβω ότι προσωπικά εγώ θα ήθελα όλες οι χώρες να έχουν ένα αντίστοιχο σύστημα αναφορών. Κάποιες το έχουν, κάποιες όχι. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για την Ευρώπη και η Ευρώπη θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες των ε, χωρών της. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου θα ήθελαν και αυτοί να προσθέσουν κάτι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο από τους φιλοξενούμενους μας. Ο πρόεδρός σας τα είπε όλα ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ Φιλ. Ελπίζω να συναντηθούμε εκ νέου. Τώρα θα ξεκινήσουμε μετά από τη χαρά που μας έδωσε η παρουσίαση την τακτική μας εργασία. Θα περάσουμε στο 6 της ημερήσιας 6.89.98. Βρετανού υπηκόου στην Ιταλία από πλευράς ε, της Ένωσης ε, Καθηγητών, Βοηθητικών Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στην Ιταλία και επίσης η 508 και 509 όπως και η 1152. Λοιπόν, ε, ο αναφέρον είναι εδώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω. Συνειδητοποιώ ότι αποτελείστε από νέα μέλη και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ευρυτάτη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια. Σήμερα, μάλιστα, που είναι η, τα πέμπτα γενέθλια της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχω δώσει ένα ενημερωτικό σημείωμα με το ιστορικό των παραπώνων μας, των αναφορών μας και των δημοσιευμάτων του τύπου. Τον Ιανουάριο του 2011 στείλαμε μια επιστολή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελεύθερη Διακίνηση ζητώντας τους να παρέμβουν μετά από την εφαρμογή του νόμου του 2010 του γνωστού ως νόμου Τζελμίνη. Η Επιτροπή το 2014 μας είπε ότι έχει ολοκληρώσει εν πολύ στην διαδικασία αναφοράς. Ο καθηγητής μας, ο καθηγητής μάλλον Πικότη, ο δικηγόρος μας, ο οποίος έχει ε, υπερασπιστεί με επιτυχία τις δύο περιπτώσεις βοηθών καθηγητών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έστειλε μία επιστολή στις 24 Νοεμβρίου στον πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker ζητώντας ε, από την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακληθεί διότι περιλαμβάνει μία προφανή α, ουσιαστική λανθασμένη αντίληψη σε σχέση με την ερμηνεία του νόμου και θα σας το δείξω αυτό στις διαφάνειες. Αν μπορείτε παρακαλώ να βγάλετε τη διαφάνεια. Βλέπετε ότι υπάρχουν 7 στήλες. Ε, μιλάμε για, το, για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κτλ ανάλογα με τον νόμο. Θα δείτε πως οι βοηθοί καθηγητές προσελήφθησαν για πρώτη φορά το 88 με ετήσια συμβόλαια. και ε, σύμφωνα με τον νόμο ήταν συμβόλαια ορίστου χρόνου. Γι' αυτό ε, υπήρξαν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και αυτό δεν εκπλήσει κανένα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με τον Ευρωπαϊκό Νόμο γιατί ε, πρόκειται για διάκριση η οποία βασίζεται στην εθνικότητα του απασχολουμένου. Η Ιταλία λοιπόν κατήργησε τον νόμο αυτό του 80 και το 95 ψήφισε ένα νέο νόμο. Ο νόμος αυτός ήταν και αυτός ε, κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή μάλλον στάλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο αποφάσισε ότι δεν ήταν συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ιταλία λοιπόν νομοθέτησε για μια ακόμη φορά το 2004 στη στήλη 6 και αυτό έχει σημασία. Η στήλη 6 λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ο νόμος του 2004 είναι ικανός. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να τερματίζει την υπόθεσή μας και θα έπρεπε απλά οι Ιταλικές αρχές από εδώ και πέρα να κληθούν να εφαρμόσουν, αλλά δεν το έκαναν αυτό. Και δεν το έκαναν γιατί δεν έδωσαν τα, τις απαιτούμενες πιστώσεις. Συνεπώς λοιπόν οι βοηθητικοί καθηγητές επανήλθαν στο δικαστήριο για νιωστή φορά και ζήτησαν οι αμοιβέ τους να είναι συμβατές με τις συνεισφορές τους και άρχισαν να παίρνουν αποζημιώσεις και γι' αυτό ακριβώς το Ιταλικό κράτος κατέθεσε ένα νέο νόμο ε, τον Τζελμίνη ή το, στη στήλη 7. Αυτή η στήλη, αυτός ο νόμος παραβιάζει πλήρως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όπως θα δείτε από τα βέλη αποκαθιστά ουσιαστικά το νόμο του 1955 Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφυρίζει κλέφτικα Η επιστολή τώρα της Επιτροπής της 16 Ιουνίου του 2014 αγνοεί πλήρως τον νόμο 63. Τον αγνοεί πλήρως. Αγνοεί πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που σαφώς και ε, έδωσε την περιγραφή των αρχών που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Σε όλες τις εφημερίδες βλέπει σήμερα ότι το θέμα της ελεύθερης διακίνησης είναι στην επικαιρότητα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση σε όλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είτε είναι κανείς υπέρ της Ευρώπης είτε κατά της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά θέλει να ισχύει το κράτος δικαίου και να αμείβεται ο κόσμος ανάλογα με την εργασία του. Ενώ σήμερα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση τέτοια όπου μέσω της χρήσης ε, του νόμου Τζελμίνη 91 καθηγητές είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται κατά 61%. Προσέβαλαν την απόφαση αυτή, τα δικαστήρια στην Ιταλία τους αγνόησαν πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείτε στους ανθρώπους αυτούς που είναι θύματα ενός ε, νόμου που στοχεύει τους Ένους ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος τους. Σας ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Πέρες Φλόρες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μέλη του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή παρευρίσκεται εδώ, μάλλον παρευρέθη εδώ τον Νοέμβριο για να εξηγήσει προφορικά την θέση της. Το Νοέμβριο του 2013. Τότε ήρθαμε και εξηγήσαμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής εδώ στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου και δώσαμε στους αναφέροντες την δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δικιά τους επιχειρηματολογία. Έστειλαν την ε, απάντησή τους, εξετάσαμε τα επιχειρήματά τους και καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα. το οποίο μάλιστα το στείλαμε και γραπτό στους αναφέροντες τέλη Αυγούστου. Τρία είναι τα κύρια σημεία της ε, επιστολής του Αυγούστου. Πρώτον, όπως γνωρίζει αυτή η Επιτροπή, για να ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση, με βάση το άρθρο 358, το βάρος της απόδειξης το έχει η Επιτροπή. Δηλαδή η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι το κράτος μέλος έχει παραβιάσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. δεν συμφωνούμε με την ερμηνεία που δίνουν οι αναφέροντες στις αποφάσεις του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να είναι διαρκής η πρόσληψη μετά την ακύρωση του νόμου του 95, δηλαδή το συμβόλαιο να ε, θεωρηθεί ότι δεν διακόπηκε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ποτέ δεν είπε ότι αυτός ο νόμος, ο Ιταλικός του 95 ήταν ε, εναντίον του Ευρωπαϊκού Δικαίου, δεν συμβόταν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έλεγε ότι ορισμένα ε, Ιταλικά πανεπιστήμια ακολουθούν διοικητικέ πρακτικέ που δίνουν την εντύπωση ότι, ότι ε, ασκούν διακρίσει. Ότι οι καθηγητέ αυτοί υφίστανται ε, διακρίσει. Και αναφερόμαστε στα έξι πανεπιστήμια στα οποία, ε, για τα οποία μιλάει η απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί σε άλλα πανεπιστήμια έγιναν συλλογικέ διαπραγματεύσει και ε, συμβόλαια με βάση στις διαπραγματεύσεις. Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι μετά το 1995 θα έπρεπε να εφαρμοστούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κράτους ε, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό είναι μια, ένα από τα επιχειρήματα της αίτησης. Η εξομοίωση των Λετόρι με το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι επίσης ένα από τα επιχειρήματα των, ε, ε, των ετούντων και πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια εξομοίωση. Αυτό που δέχθηκε το δικαστήριο είναι ότι οι Λετόροι θα μπορούσαν να μεταβληθεί η σχέση εργασία τους και να περάσουν στην κατηγορία των βοηθών. Αναζητώ τη λέξη στα Ιταλικά κολαμπορατόρια, experti linguistici. Ε, πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία, δεν πρόκειται για διδακτικό προσωπικό. Επομένως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έλαβε θέση από αυτού που να δίνει δικαίω στους προσφέροντες και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία δεν είχε δικαίωμα να πράξει όπως έπραξε. Γι' αυτό το λόγο, μετά από τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, λαμβάνοντα υπόψη τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 45. Και το Τρίτο ζήτημα είναι η παράταση στις περιπτώσεις που βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίων. Η παράταση του συμβολίου. Με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 3 του, νόμου Τζελμίνη, βάση του οποίου ε, όλες οι υποθέσεις οι οποίες βρισκόντουσαν ενώπιον των δικαστηρίων αυτομάτως θεωρούνταν λήξασες, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, μάλλον, το ζήτημα είναι να υπάρξει ορθή διαδικασία και αποζημίωση. Οι ετούντες πιστεύουν ότι αυτό δεν ισχύει και επικαλούνται τον χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι με βάση μάλλον τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 της χάρτας δεν είναι απόλυτα αλλά μπορούν να ε, υφίστανται περιορισμούς σταθμίζοντας τις ε, προϋποθέσεις του άρθρου 52 ε, παράγραφος 1, δηλαδή να προβλέπεται από νόμο, να δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφυγής και επίσης να υπάρχει σεβασμός της αναλογικότητας στην προσπάθεια εξυπηρέτησης του γενικού συμφερόντος. Γενικού συμφερόντος. η Επιτροπή δεν θα ήθελε να επέμβει σε μια διαδικασία αστικής διαφοράς Χρειάζεται να εξεταστεί. Εάν αυτή η τελευταία διάταξη του νόμου Τζερμίνη ε, είναι συμβατή με την προσπάθεια προάσπισης του γενικού συμφέροντος και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τον ε, νόμο Τζερμίνη με βάση το άρθρο 52 της ΧΑΠΤΑΣ Και θα ενημερώσουμε την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Την Παρασκευή, πριν το Σαββατοκύριακο, μόλις, λάβαμε στα αγγλικά μονάχα το, ένα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις της Επιτροπής, αυτό που μόλις μας είπατε. Τώρα σας δίνω το λόγο πάλι στον Ετούντα. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή αναφέρεται και παραθέτει την απόφαση του δικαστηρίου που βρίσκεται στην ε, στήλη 7 του χαρτιού που σας έδωσε, του που σας μοιράσα. Αναφέρεστε σε αυτή την απόφαση. Αλλά την ερμηνεύετε λανθασμένα. Λέτε ότι ο... το δικαστήριο εξέτασε μόνο τον νόμο του 2010 και τον νόμο του 1995, ενώ στην πραγματικότητα εξέτασε τον νόμο του 4, 2004. Πώς μπορεί να αγνοεί η Επιτροπή ότι η τελευταία απόφαση του δικαστηρίου πώς μπορεί να την αγνοεί πλήρως στην ανάλυση της. Είμαι σίγουρος ότι κανένας σε αυτή την αίθουσα δεν κατάλαβε ακριβώς τι είπε η Επιτροπή, γιατί η ίδια η Επιτροπή πιστεύω έχει, βρίσκεται σε σύγχυση και δεν έχει απαντήσει στην, στο βασικό ερώτημα, το οποίο σας παρακαλώ τώρα να απαντήσετε με βάση τον νόμο Τζελμίνη 91 εργαζόμενοι μη Ιταλοί και μόνο μη Ιταλοί ε, υπέστησαν μείωση μισθού χωρί να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε δικαστήριο για να αποζημιωθούν για αυτό. Και τώρα μου λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα θεωρήσει ότι αυτό είναι προβληματικό, ότι είναι ξεκάθαρη ε, διακριτική μεταχείριση με βάση την εθνικότητα. Θέλετε να απαντήσετε, η Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Δεν μπορώ να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το νόμο Τζελμίνη και ειδικά τις περιπτώσεις που απορρίφθηκαν. Εξετάζουμε λοιπόν το νόμο αυτό, άρθρο 47 και θα επανέλθουμε στην Επιτροπή και σε εσά όταν έχουμε ολοκληρώσει τον ενδελεχή μας έλεγχο. Η Πρόεδρος, έξοχα, ο Um, κυρία θα ήθελα να πω ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης ε, διακίνησης εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μη επιβολή διακρίσεων λόγω ηθαγένειας. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν ε, ε, στόχευθεί λέκτορες, οι διδάσκοντες λόγω της ηθαγένειάς τους. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανισχυτική η απάντηση της ε, Κομισιόν ε, του Αυγούστου και έχω, έχει αυξηθεί η ανησυχία μου περαιτέρω σήμερα διότι ένα, μία πτυχή ε, της αναφοράς αυτής ε, και της υπόθεσης γενικά αφορά την απαγόρευση προσφυγής στα δικαστήρια ή την έλλειψη μάλλον δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια. Ε, τώρα, αλλοδαποί εργαζόμενοι στην Ιταλία δεν έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να μην ερμηνευτεί ως διάκριση εναντίον τους. Η Κομισιόν λοιπόν έχει κλείσει το, το φάκελο ενός τμήματος της αναφοράς αλλά έχει μείνει ανοιχτό ένα άλλο μέρος το οποίο είναι ακόμα εξετάζει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτός ολόκληρος το φάκελο της αναφοράς διότι αναμένουμε από την τελική κυβέρνηση μία ε, δικαιολογημένη, δικαιολογημένη γνωμοδότηση rights e Τεκμηριωμένη γνωμοδότηση επί της υποθέσεως για να δούμε τι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στο εθνικό επίπεδο. Και ε, υπάρχουν πραγματικά βάσιμες θεμελιώδεις ανησυχίες και αντιρρήσεις σε μια τέτοιου είδους τεκμηρίωση ε, από την πλευρά κομισιών. Διότι εδώ διακυβεύεται και στρεβλώνεται η κοινωνική πτυχή ε, της, του καταστατικού του, του, χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, του, είναι θεμελιώδης αρχή αυτή η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή και από την Ιταλική κυβέρνηση και θα παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη της υποθέσεως. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Υπάρχει άλλο μέλος που θέλει... Ο κύριος Βαλέντσα θέλει να παρέμβει. Ειλικρινά, κυρία Πρόεδρε, ήρθα εδώ ελπίζοντας ότι θα κλείσει αυτός ο φάκελος. Έχει ξεκινήσει. Πότε έγινε η πρώτη αναφορά, το 98. Ε, πάρα πολύ έχει τραβήξει. Όμως, φαίνεται ότι δεν έχει μελετήσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, σωστά, και ο νόμος ο νόμος του Τζελμίνη του 2010 ε, μας ε, πιέζει να επανεξετάσουμε ολόκληρο το θέμα. Παρακολούθησα την, όσα είπε ο αναφέρον και αυτά που κατάλαβα είναι ότι αντιτίθενται ριζικά σε αυτά που είπε η Κομισιόν τελικά δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ολοκληρώσει την μελέτη της για να μας παρουσιάσει μία τεκμηρωμένη άποψη για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πριν έχουμε την πλήρη και τελική αξιολόγηση της Κομισιόν δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Η Πρόεδρος, η τελευταία πρόταση της παρέμβασης της Κομισιόν είπε μόλις αυτή η συγκεκριμένη ενημέρωση, η πληροφόρηση υπάρχει για τις επιπτώσεις των αποφάσεων ε, του νόμου, του περιεχομένου του νόμου αυτού και μόλις αυτές οι πληροφορίες ε, έχουν ληφθεί από την Ιταλική κυβέρνηση η Κομισιόν θα αξιολογήσει ε, αυτή την, τις επιπτώσεις και θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα στην Επιτροπή μας. Εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες ε, των προλαλήσαντων διότι δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεδομένου ότι την απάντησή της η Κομισιόν μας την έδωσε την Παρασκευή πριν από το Σαββατοκύριακο για να συζητηθεί τη Δευτέρα. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ε, είναι μία ε, εκρεμή υπόθεση από το 1998 Τρεις φορές έχει γίνει, έξι με διορθώνουν, έξι έχει, φορές έχει γίνει προσφυγή στο ΔΕΚ. Ε, ε, αυτό είναι φοβερό, φοβερό. Και ε, το, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το αρμόδιο όργανο για την ερμηνεία του νόμου και η Κομισιόν πρέπει να συμμορφωθεί, να αντιδράσει, μάλλον να ανταποκριθεί. Ε, δεν θα ήθελα να σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι, αλλά για να είμαι ευγενική, σας ρωτώ, θα έχετε ολοκληρώσει μέχρι τον Ιανουάριο πλήρως την αξιολόγηση του άρθρου 47 του νόμου Τζελμίνη. Μπορούμε να αναμείνουμε από εσά αυτή τη δέσμευση. Και θα σας βοηθούσε εάν εμείς από την Επιτροπή Αναφορών στείλουμε μία επιστολή μας στις Ιταλικές Αρχές ε, που να λέει ξεκάθαρα ότι είμαστε εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν που είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσει αυτό το θέμα το οποίο είναι, ντροπιάζει και εξέτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα. Η Κομισιόν Βεβαίω, έχετε το δικαίωμα αυτό και ίσως έτσι μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση ε, για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της έρευνας. Ωραία. Λέει η πρόεδρος, η αναφορά μένει πλήρως ε, ανοιχτή, ο φάκελος μένει ανοιχτός, ε, θα αποτανθούμε στην αρμόδια αρχή και αναμένουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από πλευράς Κομισιόν εντός ενός μηνός. Μπορούμε το Αναμένουμε αυτό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Πολύ ωραία, έξοχα. Α, παρεμβαίνει η Κομισιόν. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ αυτό, διότι αυτό αξιολογείται, ε, μελετάται και από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, η οποία δεν είναι παρούσα σήμερα. Δεν μπορώ λοιπόν συγκεκριμένα να δεσμευτώ επί του χρονοδιογράμματος. Η Πρόεδρος, έπρεπε να είναι εδώ εκπρόσωπος της ε, DG Justice ε, έπρεπε να είναι, είχαν, τους είχαμε ζητήσει να έρθουν πολύ λυπάμαι λέει η πρόεδρος, συνήθως δεν είμαι τόσο αυστηρή εμείς στη Σουηδία έχουμε, έχουμε ψύχρεμο είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι εκεί στο βορρά αλλά έχω λίγο ανάψει τώρα λέει η πρόεδρος η Κομισιόν Κοιτάξτε, ναι, ναι, ε, θα, θα τους ζητήσω να επανέλθουν το ταχύτερο. Ας πούμε, θα, ζητήσω να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τους ε, συνεργάτες μου το ταχύτερο. Ωραία λέει η πρόεδρος. Ας πούμε σε ένα μήνα. Λοιπόν, πίεση σε εσά, εσεί τι υπηρεσίε σα και θα στείλουμε επιστολή στι Ιταλικέ Αρχέ, ώστε μαζί, συνεργαζόμενοι, να μπορέσουμε επιτέλου να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία. Ε, τώρα θα δώσω πάλι το λόγο στην Κομισιόν κατευθείαν για τις αναφορές 508 και 509 εφόσον οι αναφέροντες λείπουν, δεν είναι παρόντες. Έχετε τίποτα να μας πείτε, είναι το ίδιο θέμα, είναι αυτή η διακριτική μεταχείριση των δασκάλων ξένων γλωσσών ε, στα Ιταλικά Πανεπιστήμια. Λίγο πολύ παρόμοιο θέμα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα εκτός από αυτά τα οποία η συνάδελφός μας κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ ετώνησε ότι δεν θα πρέπει, θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι δεν δημιουργούνται διακριτικές επιπτώσεις. Προχωρούμε στο θέμα 7. Αναφορά 1169 του 2013 έχει 135 υπογραφές, αφορά την εργασιακή ανασφάλεια στα Ιταλικά σχολεία και απευθύνουμε κατευθείαν στην Κομισιόν ή ο Σάσα Γκάρμπεν ή ο Τιμ Ρέντροπ θα μας μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η αναφορά αυτή πράγματι αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά την αναγνώριση ορισμένων ικανοτήτων διδασκαλίας και διπλωμάτων και το άλλο αφορά μόνιμη, στο μόνιμο χαρακτήρα της συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης. Για το πρώτο θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχθεί ε, αναφορές και παράπονα και για αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις. Ήρθαμε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Αγορών λόγω της ύπαρξης της οδηγίας αναγνώρισης διπλωμάτων. Η ουσία είναι ότι ε, η αναγνώριση των Ιταλικών διπλωμάτων είναι μια καθαρός εθνική κατάσταση και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση κοινοτική αρμοδιότητα, δεν υπάρχει η διαμεθοριακή επίπτωση, δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, συνεπώς το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά επί τη βάση του Ιταλικού νόμου. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος για να παρέμβει κανείς στην συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν υπάρχει διαμεθοριακή επίπτωση. Για το δεύτερο θέμα τώρα, τη μονιμότητα της μορφής απασχόλησης, τα αγαπητά μέλη θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές οδηγίες οι οποίες ασχολούνται με το θέμα αυτό και έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει μια διαδικασία επιπαραβάση η οποία είναι εν εξελίξη εις βάρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε και μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε προκαταρκτικό επίπεδο η λεγόμενη απόφαση Μάσκολο. Ε, και την Πέμπτη θα συναντηθούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια αντιπροσωπεία της Ιταλικής, ε, του Ιταλικού Δημοσίου για να συζητήσουμε το θέμα των διαδικασιών επί και τις αποφάσεις επιπτώσεις μάλλον ε, της δικαστικής απόφασης για την αυξημένη χρήση εξωτερικών συνεργατών στα Ιταλικά σχολεία. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Ο κύριος Βαλέντσα είναι σαφές ότι η Ιταλία θα πρέπει να σεβαστεί το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας για μόνιμη απασχόληση. Οι Ιταλικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Δεν μπορούμε βέβαια εμείς να υποστηρίξουμε την συνεχή ανανόηση αυτών των ορισμένου χρόνου μορφών απασχόλησης. Το θέμα λοιπόν είναι να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα αυτό οι Ιταλοί και το θέμα είναι αν θα την κρατήσουμε ανοιχτή ή όχι. Αν υπάρχουν καταχρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κυρώσεις εις βάρος αυτών που το κάνουν αλλά πέραν αυτού τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε θετικά. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Ελεονόρα. Εγώ απλά λαμβάνω υπόψη την περιγραφή της κατάστασης, μια σοβαρή κατάσταση. Απαιτείται εδώ για να μπορέσουμε εμείς να εντοπίσουμε τις σωστές πρακτικές ε, χρειάζεται μερικές φορές να εντοπίσουμε και τα λάθη μας και να μας πούνε ποια είναι τα λάθη μας. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι μια ιστορική απόφαση. Σύνεπως θα πρέπει μέσω αυτής να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να αντιμετωπίσουμε την τραγική κατάσταση της ε, προσωρινής απασχόλησης στα δημόσια Ιταλικά σχολεία. Η κατάσταση αυτή νομίζω ότι στην ουσία προκαλεί βλάβη στην οικονομία της χώρας, μια χώρα η οποία οικονομικά είναι ιδιαίτερο εύθραστη. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά και θα πρέπει επίσης να πιέσουμε έτσι ώστε οι Ιταλικές αρχές να πάρουν πιο συγκεκριμένες και πιο σοβαρές αποφάσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ε, ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις δύο επιπλέον υποθέσεις οι οποίες είναι σε δικαστική εκκρεμότητα, σε δικαστική διαδικασία. Ε, βασικά διαπιστώνεται εδώ ότι υπάρχει αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει ε, όταν μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για τη στάση των Ιταλικών αρχών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλες αναφορές οι οποίες αφορούν το θέμα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορούμε να τις βάλουμε όλες μαζί. Βέβαια ε, υπάρχει μια διαφορά εδώ σε σχέση με τα απαιτούμενα επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα συνδέσουμε ή να μην τα συνδέσουμε. Πάντως ε, η ουσία είναι ανοιχτή σε σχέση και με τις δύο άλλες αναφορές οι οποίες δεν εκκρεμούν σήμερα. Εγώ θα εκτιμούσα παρακαλώ να τις ομαδοποιήσετε και ό,τι συνδέεται, ό,τι προσωμιάζει εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο ουσίας θα πρέπει να ομαδοποιείται και να αντιμετωπιστούν από κοινού. Εφόσον λοιπόν λάβετε περισσότερες πληροφορίες τότε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό θα ήταν το πιο νομίζω σωστό. Σας ευχαριστώ. Καλώς λοιπόν συνεχίζουμε στο 8. Πρόκειται για την ε, 1961 του Εύδοτ Μάρνελ εξ ονόματος των απεργών της Κάμελ Λέιρντ. Ο κύριος Μαρνέλ έχει το λόγο. Του δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των απεργών του, ε, απεργίε του 1984 στα ναυπηγεία Καμελέιτ, θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας σήμερα για να σας παρουσιάσω την αναφορά μας προσωπικά. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή στην προσπάθεια που ε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια για να αποκαταστήσουμε την αδικία που έγινε εναντίον μας. Από το 1984 συστηματικά έχουμε προσπαθήσει να αποκτήσουμε πληροφορίες, να βρούμε απαντήσεις, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επανορθωθεί αυτή η σοβαρή παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. Δεν, έχουμε τη δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες και ε, να βρούμε τα πατούμενα τεκμήρια που θα μας βοηθούσαν στην παρουσίαση της υπόθεσή μας. Έτσι λοιπόν απευθυνόμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχοντας πλέον εξαντλήσει όλα τα άλλα νομικά ε, μέσα στη διάθεσή μας στο εθνικό επίπεδο. Και ελπίζω ότι τουλάχιστον έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Να σας δώσω λίγο το ιστορικό της υπόθεσης. Τον Μάιο του 1984 η Κάμελ Λέατ, που τότε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά ναυπηγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε υποχρεωτικές απολύσεις ε, του 50% του εργατικού δυναμικού τους. Στο Λίβερπουλ, σε μια περιοχή η οποία είχε ήδη πολύ υψηλή ανεργία. Γνωρίζαμε ότι ο στόχος τη διοίκησης ήταν να κλείσει τα ναυπηγεία παράλληλο που το αρνείτο ε, προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, αλλά ε, απέτυχε αυτή η προσπάθεια και ξεκίνησε απεργία, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις εργασίες μας. Εκείνη την εποχή, ας μην ξεχνούμε ότι η κυβέρνηση ήταν ε, η κυβέρνηση της Μάρκαρετ Θάτσερ, η οποία ήταν γενικότερα εναντίον των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και μιλάμε επίσης για την περίοδο της μεγάλης απεργίας των ανθρακορίχων τον Ιούνιο του 1984 στο ναυπηγείο εκείνη την εποχή υπήρχε μια πλατφόρμα εξόριξης φυσικού αερίου και μια φρεγάτα του βασιλικού ναυτικού την οποία ε, κατέλαβαν 40 ε, εργαζόμενοι. Τέτοιου τύπου ενέργειες ήταν συνήθεις στις απεργίες εκείνη την εποχή. Στις 3 Σεπτεμβρίου απολυθήκαμε εξαιτίας ε, απαράδεκτης συμπεριφοράς και αυτό όχι μόνο οι καταληψίες αλλά επίσης και δύο μακριθυντευόμενοι οι οποίοι υποστήριζαν τους απεργούς. Από τότε ένας από αυτούς έχει αποβιώσει. Στις 5 Σεπτεμβρίου μας, έδωσε, ε, μας κοινοποιήθηκε η εντολή να φύγουμε από την, το ναυπηγείο. Εκδικάστηκε η απόθεση μας Ρήμιν κάτι που θεωρούμε ότι ήταν μια δυσανάλογη ε, αντίδραση στο νόμιμο μας δικαίωμα στην απεργία. Οκτωβρίου Πολλοί από τους απεργούς συνελήφθησαν εντός των αυπηγείων. Στις 3 Οκτωβρίου ε, ένας ε, αστυνομικός με πολιτικά, του οποίου την ταυτότητα αγνοούμε, μας έδωσε την εντολή να φύγουμε αμέσως από τα δύο σκάφη, γιατί διαφορετικά θα κινδύνευε η ζωή μας. Την ίδια στιγμή βλέπαμε κομμάντος από τις ε, ειδικέ δυνάμεις να σκαρφαλώνουν σε έναν πύργο εκεί κοντά. Δεν θέλαμε προφανώς να κινδυνεύσει κανένας και ε, αμέσως απομακρυνθήκαμε. Ε, οι απεργοί συνελήφθησαν, τους πέρασαν χειροπέδες και ε, τους έστειλαν στη φυλακή Walton, που μια φυλακή ε, υψίστης ασφαλείας. είναι σημαντικό να σημειώσουμε κατά τη διάρκεια της κατάληψης περνούσαμε κάθε πρωί μπροστά από τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν μας είχαν πει τίποτα έως τότε ότι παρανομούμε για παράδειγμα. Επί τέσσερις εβδομάδες οι συλληφθέντες απεργοί υποστήκαμε ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείριση βρισκόμασταν ε, κρατούμενοι σε απομόνωση μέχρι και 23 ώρες την ημέρα χωρίς επαφή με τον εξωκόσμο στην ε, πτέρυγα υψής της ασφαλείας αυτής της φυλακής. Αυτό είναι προφανέστατα μια δυσανάλογη αντίδραση στο νόμιμο, στην άσκηση του νόμιμου δικαιώματο μα στην απεργία. Μια απεργία η οποία έληξε ειρηνικά και χωρίς καμία ζημιά στι περιουσίε των ναυπηγείων. Ποτέ δεν μπορέσαμε από τότε να βρούμε τα στοιχεία, τα, τα έγγραφα μιας απόφασης δικαστικής που να δικαιολογεί αυτή την κράτηση. Ε, χάσαμε τα δικαιώματά μας στην αποζημίωση και στις ασφαλιστικές μας εισφορές και από τότε κανένας από τους απεργούς δεν μπόρεσε να βρει δουλειά στον κλάδο. Στην πραγματικότητα μπήκαμε στη μαύρη λίστα εξαιτία του ε, δράσεως μας της ε, συνδικαλιστικής. προσφύγαμε στα δικαστήρια ως, για να κηρυχθεί η απόλυσή μας παράνομη αλλά το εργατοδικείο απέρριψε αυτές τις προσφυγές και δεν είχαμε δικαίωμα έφεσης. Δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο, κανένα έγγραφο που να συνδέεται με αυτές τις αποφάσεις. Μας φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Έχουμε προσπαθήσει να αξιοποιήσουμε ε, την νομοθεσία για την πρόσβαση, την δημόσια πρόσβαση στα κρατικά έγγραφα. Την τελευταία προσπάθεια έγινε το 2012 ε, έχουμε απευθυνθεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά ποτέ δεν μας δόθηκε μια ικανοποιητική απάντηση και κανείς δεν μας έχει εξηγήσει γιατί αυτά τα έγγραφα δεν βρίσκονται πουθενά. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι μια φυσιολογική ε, ε, λειτουργία της διοικητικής μηχανής ούτε του κράτους, ούτε της αστυνομίας, ούτε της δικαστικής εξουσίας. Μετά τον θάνατο της Μάργαρετ Θάτσερ, αποκαλύφθηκαν διάφορα εμπιστευτικά σημειώματα που είχαν συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και φαίνεται ότι ήδη από τις 19 Ιουλίου του 1984 είχε συζητηθεί στο Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο η πιθανότητα να κλείσει το ναυπηγείο. Κάτι το οποίο ε, αρνεί το η του ναυπηγείου από τότε. Γιατί λοιπόν προσφεύγουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά μας, την ελευθερία, στη δημοκρατία, στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως ε, ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η έντιμη δίκη, η πρόσβασή μας σε μια αναλογική και δίκαιη δικαστική διαδικασία, η πρόσβασή μας σε πληροφορίες που μας αφορούν ε, και, και έχουν παραβιαστεί τα συνδικαλιστικά μα δικαιώματα. Η φυλάκιση των απεργών επίσης έγινε κατά παράβαση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα οι απεργοί τιμωρήθηκαν επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά στη συνάθρηση και το δικαίωμα συνδικαλιστικής δράση. Ποτέ μετά από αυτή την απεργία οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να βρουν δουλειά αλλού σε άλλο ναυπηγείο στον κλάδο. Στην πραγματικότητα μπήκαν σε μια βαύρη λίστα όλες αυτές οι ενέργειες, όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν με πλήρη περιφρόνηση στην ε, ορθή νομική διαδικασία και το γεγονό ότι δεν μπορέσαμε να, δεν, δεν μας έδωσε κανείς δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούσαν στην υπόθεσή μας υπονόμευσε το δικαίωμά μας σε νομική προστασία. Δεν μπορέσαμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας νομικά. Συμπερασματικά θα πω ότι ε, δυστυχώς 7 από τους απεργούς έχουν πια πεθάνει. Αλλά υπάρχουν οι οικογένειές τους που συνεχίζουν να αναζητούν δικαιοσύνη. Και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανταποκριθεί σε αυτή την αναφορά. Θα ξεκινήσει μια ε, ενδελεχή έρευνα έτσι ώστε να βρεθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα εξηγήσουν πώς ελήφθησαν αυτές οι δυσανάλογα δυσμενείς αποφάσεις που μας επηρέασαν. Ζητούμε να αναγνωριστεί αυτό το δικαστικό σφάλμα και να, μας να, να, να δοθεί επισήμως μια ε, συγνώμη και μια αποζημίωση. Σας ευχαριστώ. Πολύ συγκινητική η ιστορία σας. Πράγματι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε τα οποία συνέβησαν αυτά που είπατε και σας ευχαριστούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σάσα Γκάλμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ίδιος ο, ο αναφέρον και οι συνάδελφοί του. Οι αναφέροντες λέγουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε όλα τα θέματα τα οποία έθεσε ο αναφέρον και βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης της ανάλυσης της. Δεν έχω να πω κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Γενικότερα θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι την εποχή που γινόντουσαν αυτά τα θέματα η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είχε ακόμα διακηρυχθεί. Παρ' όλα αυτά ε, υπήρχαν ε, συγκεκριμένα δικαιώματα, τμήματα του κοινοτικού τότε δικαίου και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνουν σεβαστά από τα κράτη-μέλη. Αλλά μόνο τώρα με την ε, ισχύ του, του θεμελιώδους χάρτη ανήκουν στο συνταγματικό θα έλεγα χάρτη των κοινοτικών γιατί αλλιώς ξέρετε ότι στα πλαίσια της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν συμμετέχει ε, πλήρως στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι σε θέση να πει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν πράγματι κινήθηκε στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου και αν το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν τμήμα του κοινοτικού δικαίου ή κάτω από το κοινοτικό δίκαιο, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου. Sorry. Thank you very much. And the floor goes to my colleague, Mrs. Curtin Darling. Η κυρία Darling. Thank you very much, Chair. Um, I'd like to um, also echo your... Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μανέλ γιατί στάθηκε αρκετά γενναίος να έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μας πει τι συνέβη εδώ και 30 περίπου χρόνια. Είναι μία σειρά ιστορικών δικαστικών λανθασμένων αποφάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει ακριβώς να πούμε ότι αυτές οι αποτυχημένες αποφάσεις είχαν σαφέστατες βιωματικές συνέπειες σε αυτούς οι οποίοι είχαν εμπλακεί. Πολλοί μπήκαν σε μαυροπίνακες και δεν μπόρεσαν να εργαστούν εκ νέου στις βιομηχανίες και στο χώρο στον οποίο είχαν προσόντα με τρομερές συνέπειες. Ε, το ότι τέσσερα αδέλφια για ένα μήνα φυλακίστηκαν σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να πάνε στην κηδεία της μητέρας τους, κάτι το οποίο ποτέ δεν μπορεί γι' αυτό να αποζημιωθούν. Ε, και γενικά δεν σεβάστηκαν τότε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 30 χρόνια και έχει κάνει εκστρατείες ε, όπως και πολίτες ε, όπως ο κύριος Μανέλ έχει συγκεκριμένα και εκτιμένα δικαιώματα όπως σωστή ε, διαβούλευση και αναζήτηση στοιχείων σωστή είναι ενημέρωση, δικαιωματική γνώση στοιχείων κτλ έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάπως την κατάσταση στις συνέπειές της τουλάχιστον και να καταλάβουμε γιατί συνέβη αυτό το οποίο συνέβη εις βάρος τους. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει ε, να ζητήσουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των απλών πολιτών απέναντι στην κρατική εξουσία και κυρίως του τρόπου με τον οποίο ασκείται αυτή είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τρέχει στην παρούσα φάση μία ανάλυση. Αυτό σημαίνει θα ακούσουμε σε κάποια φάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. Αλλά νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει την Βρετανική κυβέρνηση και να ελέγξει την κατάσταση και να μας ενημερώσει και τι γνωρίζει και τι στοιχεία μπορεί ακόμα και σήμερα να ευρεθούν. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα για κάτι τέτοιο. Είναι 30 χρόνια πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει ε, να υπάρξει έστω κάποιο μικρό επίπεδο απόδοσης δικαιοσύνης για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Να πούμε επίσης ότι στα κείμενα αυτά συστήνεται να ζητηθεί μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από την Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε σχέση με τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και σε σωστή ενημέρωση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε έτσι ώστε να υπάρξει μια επανόρθωση. Louise. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές στην απογευματινή συνεδρίαση ότι υπάρχουν πολλά να γίνουν στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των δικαιωμάτων που έχουν σχέση με την εργασία και τον τρόπο εργασίας. και μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην απεργία, το οποίο είναι ένα δικαίωμα πλήρως αναγνωρισμένο. Eh, Φυσικά αυτά έχουν αλλάξει στις διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια με τις διάφορες αποφάσεις και εναλλαγές κυβερνητικές και νομοθετικές αλλά δεν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει ε, περιορισμός. Λοιπόν, ε, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα και έστω και 30 χρόνια αργότερα να αποκατασταθούν τα δικαιώματα τα οποία έχουν θίξει με τόσο ε, σημαντικό τρόπο τους εργαζομένους και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην γνώση έτσι ώστε να γνωρίζει ακριβώς τι είχε συμβεί με πλήρη διαφάνεια. Από πλευράς μας λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη αναφορά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να συνεχίσει η διερεύνησή της, όπως πρότεινε και η προηγούμενη συνάδελφος. Ε, θα είναι ενδιαφέρον ιδιαίτερα από πλευράς της ΛΥΜΠΕ να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης ε, του τι μπορεί να γίνει σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των εργασιακών όπως συγκεκριμένα του δικαιώματος στην εργασία. Στην απεργία, συγγνώμη. Thank you very much. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι σε αυτή την περίπτωση συμμεριζόμαστε τις απόψεις της Κομισιόν και υπάρχει σύμπτωση απόψεων σε αυτό το θέμα. Και τώρα Ευχαριστώ, δίνω το λόγο στον κύριο Μαρνέλ, στον αναφέροντα, για την ε, τελευταία λέξη, για να έχει την τελευταία λέξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέχομαι τις παρατηρήσεις που έγινα και χαίρομαι που θα μας ε, βοηθήσετε στην επιδίωξη δικαιοσύνης. Αυτά θα μεταδώσω πίσω στην έδρα μου και ε, ενδέχεται να διαγράφεται κάποιο φως στη στενοπό κάποιο φως στο τούνελ εάν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει να βρούμε τη λύση. Ο πρόεδρος, ο κύριος το Πορέμπα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να υποστηρίξω τα επιχειρήματα της κυρίας Hilton Darling και της κυρίας Ρούιθ τα επιχειρήματά τους. Αναγνωρίζω τα δικαιώματα των απεργούντων, αναγνωρίζω τις ε, προσπάθειές τους, το χρόνο που διαθέτουν εις βάρος της προσωπικής τους ζωής για να υπεραμεινθούν των δικαιωμάτων των εργαζομένων και που πολλές φορές αδικούνται ή υφίστανται σοβαρές παρενοχλήσεις και υποστηρίζω πλήρως την πρόταση να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση, ο φάκελος. Η πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε μία ε, ομόφωνη άποψη, ε, ένα κονσένσους στην Επιτροπή Αναφορών. Αναγνωρίζουμε ότι εδώ διεπράχθη μία σοβαρή αδικία, η οποία είχε σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των, ενδιαφερ... των Περιμένουμε μία ε, ε, αξιολόγηση της ε, νομολογίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διότι χρειάζεται μία ερμηνεία τελεσίδικη και αυτό το που θέλω να τονίσω είναι ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάθε ένα θυγόμενο και το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν είναι να ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοιχτός και ε, ε, παράλληλα με την εργασία της Κομισιόν η Επιτροπή μας η Επιτροπή Αναφορών θα στείλει μία επιστολή στις αρχές του Ηνημένου Βασιλείου ζητώντας μία επίσημη συγγνώμη ε, για την αδικία που διαπράχθη. Αποζημίωση δεν νομίζω να μπορεί να ζητηθεί αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ε, δίκαιο μήνυμα ε, θα σταλεί στους στιγόμενους με αυτή την επίσημη επιστολή αναγνώρισης αδικίας και συγγνώμης. Πολύ ωραία έξοχα. Ε, συνεχίζουμε τώρα με το θέμα 9 που είναι η αναφορά του Ραφάλ Νταμπρόφσκι για την ε, κατασκευή του οδικού άξονα Βία Καρπάθια, Πολωνία, Λιθουανία, Σλοβακία. Από την Πολωνία πιστεύω θα καταλήξει αν δεν κάνω λάθος η Θεσσαλονίκη αυτός ο άξονας. Ο κύριος Τόμας Πορέμπα είναι μαζί μας για να... Εσείς είσαστε ακριβώς. Είσαστε λοιπόν εδώ εκπροσωπώντας τον κύριο Νταμπρόφσκι και επίσης ο κύριος Κάσπριτς και λυπάμαι αν δεν προφέρω απολύτως σωστά το όνομά σας είναι ο σύμβουλος στα αρμόδια θέματα στην μόνιμη επιτροπή της μόνιμη αντιπροσωπεία Πολωνίας ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και τους δύο λοιπόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μπορέμπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα, ήθελα να ε, μιλήσω στα πολωνικά ε, για να είμαι ακριβής και να μπορώ ακριβώς να ε, εξηγήσω με ακρίβεια και να γίνω κατανοητός από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Συνεχίζω λοιπόν στα πολωνικά. Είναι η δεύτερη φορά ε, που η Επιτροπή Αναφορών συζητεί αυτό τον οδικό άξονα, Βία Καρπάσια. Όπως ανέφερε η κυρία Πρόεδρος. Ο άξονας αυτός ε, περνάει από την ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Λιθουανία μέσω Πολωνίας, Σλοβακίας ε, και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια, ένας πάρα πολύ σημαντικός οδικός άξονας που εάν είχε εξυγχρονιστεί ε, και όταν θα εξυγχρονιστεί και βελτιωθεί ε, θα συνεισφέρει πολύ σημαντικά στην καλύτερη και πιο βελτιωμένη πρόσβαση των ε, ε, χωρών αυτών και θα ανταποκριθεί στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία της ανάπτυξης των επικοινωνιών, των μεταφορών αλλά και στην προσφορά μεγαλύτερων ευκαιριών ανάπτυξης μέσα στην Ένωση και εκτός τούτου θα βελτιώσει και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών διότι θα προσφέρει όπως είπαμε μία καλύτερη πρόσβαση στην ανατολική πλευρά ε, της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό. Τον Απρίλιο φέτος συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η προηγούμενη Επιτροπή Μεταφορών απεφάσισε να παραμείνει ανοιχτός ο φάκελος και όπως αναφέρεται στα πρακτικά ε, προγραμματιζόταν ε, μία αποστολή παρατηρητών στην Πολωνία που θα επισκεπτόταν τα βασικά κομβικά σημεία ε, κατασκευής αυτού του οδικού άξονα για να συζητήσει τα υπάρχοντα θέματα συντομία θέλω να σας ζητήσω σήμερα να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να γίνουν σεβαστές και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την προηγούμενη Επιτροπή Αναφορών της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου έτσι ώστε αυτός ο δικός άξονας να αξιολογηθεί βάσει των συμπερασμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης. Είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος ο άξονας αυτός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω αυτό σαφέστατα, είναι στρατηγική σημασίας δεδομένο ότι θα δώσει καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης, θα βελτιώσει τις μεταφορές σε μια περιφερειακή ακραία περιοχή της Ευρωπαϊκής Υπήρου και αυτά ε, είχα να πω γενικά και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ε, συζήτηση επί του θέματος. Και τώρα το λόγο έχει η Κομισιόν. Ο κύριος Σβίνσκι. Ευχαριστώ, αξιόλογα μέλη. Μπορώ να πω ότι η Δία Καρπάσια είναι μέρος του δικτύου 10T Network, του δικτύου 10 και έχει περιληφθεί στο δίκτυο 10T ακριβώς ο άξονας αυτός από το βορρά ε, στο νότο διαμέσου της Πολωνίας. Εν συνεχεία τα διάφορα τμήματα μεταξύ Λουμπλίν και Κόσιτσε, ε, παρακάτω προς ε, Ντέμπρετσεν και λοιπά, προς την Σλοβακία και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Το δίκτυο αυτό, TEN-T, έχει ε, μελετηθεί με απόλυτη διαφάνεια, έχει συζητηθεί σε βάθος και έχει έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες αποφάσεις ε, κατασκευής του ε, οδικού άξονα που είναι μέρος του 10T, 10TAF taf Όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του άξονα, το βασικό βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την χρηματοδότηση μεταφορικών επενδύσεων είναι η Euro, το Euro Facility, το Connecting Euro Facility και ε, μέσω αυτού θα χρηματοδοτηθεί αυτός ο άξονας. Υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του οδικού δικτύου και δεδομένου ότι δίνονται χρηματοδοτήσεις και από το Ταμείο Συνοχής ε, μπορεί αυτή τη στιγμή να εμπέσει στη συγχρηματοδότηση και, του ταμείου, και από το Ταμείο Συνοχής η Βία Καρπάθια. Από την πλευρά μας λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν θεωρούμε το ένα τμήμα του δικτύου TEN πιο σημαντικό από ένα άλλο τμήμα. Τα διαχειριζόμαστε ως ισότιμα. Ε, έχουν επίσης εγκριθεί και οι νομικές πτυχές από τους νομοθέτες, ε, το, η νομική βάση ε, και όλες οι νομικές πτυχές που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Υπάρχει μόνο μία μικρή εκκριμότητα στο βορειότερο τμήμα κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας που είναι άπτεται του Βαλτικού διαδρόμου και της Βορείου θαλάσσης. Ε, η πρόεδρος. Και τώρα ανοίγουμε, ε, μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση ο κ. Βαλένσα. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση αυτή η αναφορά γιατί είναι πολιτικά φορτισμένη. Το ότι ένας συνάδελφος παρουσιάζει την αναφορά αυτή αποδεικνύει ότι είναι πολιτικά εμφόρτη και νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε σχέση με το Δία Καρπάτια. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο επίσης και για τον προϋπολογισμό του 2014 και είχαμε πει ε, τότε ότι είναι σαφής ε, η θέση της Επιτροπής ο προγραμματισμός και οι άδειε οι οποίες ζητούνται στα κράτη-μέλη είναι θέμα του Πολωνικού Υπουργείου Μεταφορών. Παρακαλώ να ζητήσω από τη γραμματεία στην παρούσα φάση να σταματήσει. Παρακαλώ ησυχία. Ε, κύριε Χατζηγεωργίου, κυρία Σακοράφα, αν μπορείτε λίγη ησυχία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ακούνε τους ε, συναδέλφους όταν η γραμματεία συζητά με άλλους συναδέλφους. Συγγνώμη κύριε Βαλένσα, απαιτείται μία κάποια τάξη. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτά τα οποία έλεγα. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω να κλείσει η αναφορά, γιατί έχει ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έγκυται στη διακριτική ευχέρεια του Πολωνικού Υπουργείου Μεταφορών να δεχθεί τις άδειες για βελτιώσεις του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Αυτό έχει υποθεί και από την κυρία Βινκόφσκα η οποία είναι σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε πλήρως τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε σχέση με αυτόν τον οδικό άξονα. Είναι σαφής η θέση της πολωνικής κυβέρνησης. Το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο διανεμήθη στα μέλη σήμερα δείχνει ότι ο κανονισμός των TEN-T ε, εδράζεται σε μια σαφέστατη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε και εμπλουτίστηκε από το 2009 ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ε, υπόλοιπους εμπλεκομένους. Τα νέα TEN-T έχουν στόχο τα λεγόμενα σύνολα δίκτυα και τα λεγόμενα κομβικά δίκτυα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των διαδικασιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν θεώρησε ότι πρέπει να λάβει υπόψη της ε, την Βία Καρπάτια γιατί ούτε τα κεφάλαια που απαιτήθηκαν ούτε οι θέσει των αστικών περιοχών τις οποίες εξυπηρετεί ε, δεν το ζήτησαν αυτό. Συνεπώς λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τελικά από μακρότατες διαδικασίες η Πολωνίδα Υπουργός Μεταφορών κάποια τμήματα τα ενέταξε στο συγκεκριμένο TNT ανάμεσα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της πολωνικής επικράτειας στον λεγόμενο διάδρομο TNT. Τώρα για τη σύνδεση Μπιάλι στο Κλούμπλιν και Ζέτσου στα σλοβακικά ε, σύνορα και αυτό συμπεριλήφθη στο πακέτο μετά από μακρότατες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η σύνδεση Μπιάλιστοκ Αυγούστους δεν περιλαμβάνεται λόγω κάποιων περιβαλλοντικών αναστολών, αν θέλετε, μέσω δηλαδή περιοχών Natura 2000, ως εκ τούτου σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψής τους. Το Βία Καρπάτια λοιπόν ή Βία Καρπάτια είναι ένα σημαντικό τμήμα του διαδρόμου ανάμεσα στον βορρά της Ευρώπης και τη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί σε επίπεδο γενικής κατεύθυνσης και γεωγραφικής τοποθέτησης αλλά όχι σε επίπεδο λεπτομεριών σε σχέση δηλαδή με τα τμήματα των οδικών δικτύων τα οποία θα εντάξουν στον διάδρομο αυτό. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, ο προϋπολογισμός του Connecting Europe που θα χρηματοδοτήσει τα TNT είναι ανεπαρκής σε σχέση με τις απαιτούμενες επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχει κρίσιμη σημασία οι διαθέσιμες πιστώσεις να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και να βελτιστοποιηθεί ο στόχος χρήσης τους. Ο διάδρομος αυτός, Βία Καρπάτια, μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί και από το Ταμείο Συνοχής όχι τα παλιότερα τμήματα του δικτύου. Το ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν τα παλιά δίκτυα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εγκαταληφθεί. Η σύστασή μου για μια ακόμη φορά λοιπόν είναι να κλείσει η αναφορά διαπαντός. Σε ευχαριστώ πολύ. Σάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, το θέμα μας είναι διπρόσωπο αυτή τη στιγμή, λέει ο μιλητής. Συμφωνώ ότι είναι εξαιρετικό, εξαιρετική σημασία ο, ο άξονας αυτός για ολόκληρη την περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτός τούτου θα υπάρχουν και διακλαδώσεις από, την, από Ανατολάς προς Δυσμάς. Και ε, ένας οδικός άξονας που θα ενώνει το βορρά με το νότο ε, είναι προφανές ότι έχει εξαιρετική σημασία. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη. Αυτό είναι το ένα πρόσωπο, μία πτυχή αν θέλετε. Τώρα έρχομαι στη δεύτερη πτυχή του έργου δεν ξέρω τι θα επιτύχουμε με μία ε, αποστολή ε, ενημερωτική, με μία αποστολή παρακολούθησης, εποπτείας στην Πολωνία. Τι, τι επιτροπή θα είναι αυτή, τι σόη αποστολή θα είναι αυτή, τι, τι θα κάνει στην Πολωνία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ιδέα έχει πολιτικό υπόβαθρο και δεν βλέπω το λόγο. Πιστεύω ότι ε, δεν έχει νόημα να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία αποστολής σε μια ομάδα παρατηρητών. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να κλείσει αυτός ο φάκελος. Ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ. Είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και το Connecting Europe Facility το έχω χειριστεί ως εισηγητής της Περιφερειακής Επιτροπής θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία το οποίο έχει σχέση με την Πολωνία. Στη Γερμανία γίνεται μεγάλος καυγάς ε, για τα έργα που προγραμματίζονται στη Βόρειο Ρινανία, Βεσφαλία, δίκτυα υψηλής ταχύτητος. Το ένα μέρος του κρατηδίου λέει πρέπει να κάνετε το α, το άλλο μέρος του κρατηδίου λέει πρέπει να κάνετε το β. Και ε, τα δύο τμήματα αυτά βρίσκονται στο δίκτυο των ευρωπαϊκών TEN Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ποια έργα θα δηλώσουμε ε, μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Δηλαδή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να καταλήξουν τελικά ποιο έργο θέλουν να προωθήσουν. Αφού αποφασίσουν αυτό οι αρμόδιες αρχές, τότε προχωρούμε στο πιο ψηλό επίπεδο, αφού μπορέσει η εθνική κυβέρνηση να υποβάλει τα συγκεκριμένα ε, προγράμματα τότε γίνεται, μετά γίνεται διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ δεν θέλω να, να, να αναμειχθώ στις λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς. Προφανώς ε, είναι ένα συνολικό, ένα σύνολο δίκτυο, ε, έχει διαφορετικά τμήματα μέσω διαφορετικών κρατών. Στην Πολωνία έχει, έγινε μια αξιολόγηση και υπήρχε μια απόφαση και η πολωνική κυβέρνηση από το 2011 μέχρι το 2015 είχε υποβάλει μία δέσμη έργων, προγραμμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί. Βλέποντας τώρα την κατάσταση επιτόπου και βλέποντας αυτό το βαλτικό οδικό διάδρομο ότι έχει δηλωθεί ως μελλοντικό έργο και ότι θα αναπτυχθεί εγώ ως Ευρωπαίος πρέπει να δεχτώ αυτή, ε, αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω βεβαίως ποιος αρμόδιος θα παρέμβει για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Δεδομένου ότι υπάρχουν ε, ακόμα αντικρώμενες απόψεις, ε, περιβαλλοντικά προβλήματα, το Natura 2000, παρεμβαίνουν διάφοροι παράγοντες και έτσι υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ τους πρέπει να πω ότι τελικά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του, της Πολωνίας, του, του πολωνικού κράτους να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια τα οποία δικαιούται να χρησιμοποιήσει. Εμείς ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να αναμειχθούμε ε, στο κρατικό επίπεδο ούτε νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ε, τοπική αξιολόγηση να στείλουμε δηλαδή παρατηρητές και να μας πούνε προτιμούμε αυτή τη διαδρομή και όχι αυτή τη διαδρομή. Ε, αυτό αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας, να μην αναμειχθούμε. Η Πρόεδρος, η Σολεντά τώρα. Σας ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Πρώτον, Νομίζω ότι σε όλους είναι σαφής η μεγάλη σημασία που έχει η υπόθεση αυτή και νομίζω ότι υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη συμφωνία να αναγνωρίσουμε τη σημασία του προβλήματος το οποίο έχει δημιουργηθεί και χωρίς να θελήσουμε σε καμία περίπτωση να θίξουμε την αυτονομία ή τις δυνατότητες λήψεως αποφάσεων της ε, πολωνικής κυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει τι δυνατότητες υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με τη χρήση ε, των ε, ταμείων συνοχής. Τώρα για την πολιτικοποίηση και κατά πόσο είναι εμφορτοπολιτική στο θέμα προφανώς. Ε, είναι σαφές ότι στο παρελθόν είχε υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την αναφορά αυτή. Ε, τι ακριβώς, ε, ε, πώς εξηγείται η συγκεκριμένη αυτή η διαφοροποίηση. Νομίζω πάντως ότι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται μία επίσκεψη στο συγκεκριμένο χώρο νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια των συντονιστών. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές πάρα πολλά αιτήματα ε, για τις επισκέψεις της συγκεκριμένη Επιτροπής και θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος ε, και να βρούμε μια κάποια λύση. Now, I Κοιτάξτε. Θα προσπαθήσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Κύριε Κακόψκι. Κακόψκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Με εξέπληξε το τοποθέτηση του κ. Βαλέτσα που αμφισβητεί κατά πόσο θα ήταν ε, ορθό να τεθεί αυτή η αναφορά, να αποσταλεί καν αυτή η αναφορά. Και μιλάμε για έναν έναν εκπρόσωπο μια πλούσια περιοχή τη Ευρώπη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι ανατολικότερε, πιο φτωχέ περιοχέ. Ναι, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τι ανατολικότερε πιο φτωχέ περιοχέ. Εάν αναρωτιέμαι αν γνωρίζει ότι η Πολωνία σήμερα δεν είναι η ίδια με εκείνη που ήταν πριν από 500 χρόνια. Κάποτε υπήρχε ένα ενιαίο κράτος που συμπεριλάμβανε τη σημερινή Σλοβακία, Λιθουανία, η αυτοκρατορία των Γεγελόνσκι. Αλλά μιλάμε για πριν 500 χρόνια. Σήμερα συζητάμε έναν ε, δρόμο ο οποίος θα ξεκινά από τη Βαλτική, θα περνάει από τη Σλοβακία, από τη Βουλγαρία, από την Πολωνία και θα φτάνει και στην ε, Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Δεν είναι απλώς πολωνικό με άλλα λόγια. Και ο κύριος Βαλένς αυτό τουλάχιστον θα ήθελα να το δεχτεί. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη στο Ανατολική Ευρώπη. Σε περιοχές οι οποίες είναι φτωχές, σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν οδικό δίκτυο. Αν κάποιο σήμερα θέλει να πάρει το αυτοκίνητο και να περάσει από την Πολωνία στην Ελλάδα, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να περάσει μέσω από την Τσεχία. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο ε, δρόμος, καλύτερο, καλύτερο οδικό δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη και αυτό είναι τραγικό. Ιδίως εάν σκεφτούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς υπονοώ την Ουκρανία και την κατάσταση εκεί και την απειλή που ε, αυτή αντιπροσωπεύει, η κατάσταση στην Ουκρανία αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα έπρεπε να επενδύουμε στις ανατολικές περιοχέ. Αυτό λοιπόν το έργο είναι απαραίτητο και θα έπρεπε να θεωρηθεί και να του δοθεί προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζω να εκπλήσω με την στάση του κ. Βαρένσα ε, και το γεγονό ότι είπε ότι είναι μια πολιτική επιλογή. Ναι, βέβαια είναι μια πολιτική επιλογή. Είναι μια γεωπολιτική στρατηγική επιλογή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Είναι στρατηγικού ενδιαφέροντο όχι μόνο για την Πολωνία, αλλά και για την ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει σοβαρά αυτό το έργο. Και γι' αυτό Σα ζητώ να άρετε το αίτημά σα να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Καλύτερα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Πρόκειται για το συμφέρον όχι μόνο της Πολωνίας, αλλά ολόκληρων των χωρών στην, ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης συνολικά. Ε, chciałam odpowiedzieć e, koledze, panu posłowi να απαντήσω. Πράγματι, είναι πολιτικό το θέμα και αυτή η αναφορά είναι ζήτησα να ενημερωθώ για τη χρηματοδότηση την εθνική για την Βία και μου δόθηκαν τα εξής στοιχεία. Μιλάμε για 6.554 συμβόλαια με συνολική αξία 33 δισεκατομμύρια λότι. Επομένως μιλάμε για ένα τεράστιο ε, ποσό. 19 δισεκατομμύρια σλότη θα ήταν η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Εάν κάνουμε την αναγωγή κατά κεφαλή, πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό, το δεύτερο μεγαλύτερο έργο στην Πολωνία. 2,5 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της περιοχής, επίσης 2 δισεκατομμύρια σχεδόν από το πρόγραμμα για την καινοτομία, το 28% αυτών των χρημάτων θα κατευθυνθεί στον τομέα των μεταφορών και 9 δισεκατομμύρια σλότη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της καινοτομίας. Επίσης υπάρχουν και πολλά project τα οποία αναφέρονται στην κοινωνική διάσταση αυτού του, έργου. 12% σε αυτό το σκέλος του προϋπολογισμού. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πολωνική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, με αυτή την αμέλεια που υπήρχε στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Δεν αδρανεί η πολωνική κυβέρνηση, γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να ζητήσω να κλείσει η αναφορά. Λοιπόν, δύο μέλη πήραν το λόγο και μίλησαν για πολλή ώρα και τώρα ξαναζητάνε το λόγο. Εν πάση περιπτώσει να μην ξεπεράσετε παρακαλώ το ένα λεπτό ο καθένας. κύριος Βαλένσα. Εγώ ζήτησα το λόγο, λέει ο κύριος Βαλένσα, διότι ο κύριος Βοητσεχόφσκι αναφέρθηκε σε μένα και σε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι εγώ είπα και μου επετέθη προσωπικά μη λέγοντας την αλήθεια. Το θέμα δεν είναι μεθοδολογικό συνάδελφοι, το θέμα είναι τι μπορεί να συμπεριληφθεί στο λεγόμενο κομβικό δίκτυο και τι μπορεί να συμπεριληφθεί στο λεγόμενο σύνολο δίκτυο, συνολικό δίκτυο. Λοιπόν, όταν υπάρχει έτσι και αλλιώ διάθεση πιστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τη χρήση τους. Δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Συγκεκριμένα ποσά ανήκουν σε συγκεκριμένα προγράμματα και σε συγκεκριμένα έργα. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, λέει ο κ. Πορέμπα. Ε, ξεκινώντας και με κάθε σεβασμό, Πρόεδρε, ε, δεν ξέρω σε τι αναφέρθηκε η κυρία, η κυρία Πιτέρα. Εγώ αναφέρομαι όχι γενικά στις επενδύσεις για την περιοχή Ποτκαρπάτια, αλλά ε, για τον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Κοιτάξτε κύριε Βαλένσα, είστε Πολωνός, εγώ και σας ενδιαφέρει αυτό, έχω υπερασπιστεί τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, τον συγκεκριμένο διάδρομο. Το θέμα όμως όπως είπαμε δεν αφορά μόνο την Πολωνία, είναι θέμα το οποίο αφορά και, αφορά και άλλες χώρες. Και εσείς σήμερα μας ζητάτε να κλείσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής και της δικής σας, όχι μόνο τις υπόλοιπες χώρες αλλά και στη δική σας χώρα. Ντρέπομαι λοιπόν για αυτό που συμβαίνει. Ντρέπομαι για σας, ντρέπομαι για αυτό το οποίο διεκδικείτε, για αυτό το οποίο ζητάτε. Είναι η πρώτη φορά που ένας Πολωνός βουλευτής ζητά ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα για τη χώρα μας να κλείσει, να τερματιστεί. Κοιτάξτε κύριε Πορέμπα, προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί, προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί μεταξύ μας. Αν έχετε όρεξη να τσακωθείτε, να πάτε έξω να τσακωθείτε, όχι μέσα στην αίθουσα παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Εγώ σαν Ευρωπαία πολίτης ενδιαφέρομαι. Θέλω την άποψη επίσης και τον εκπρόσωπο της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Κάσπεριτς. και διορθώνει ο κύριος Κάσπερι και λέει ότι λέγομαι Κάσπριτς. Εγώ είμαι υπάλληλο, συνεπώς δεν ανήκω στα πολιτικά κόμματα και εγώ ήμουν υπάλληλο για τα συγκεκριμένα θέματα και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την παρούσα κυβέρνηση. Ήμουν υπεύθυνο και για θέματα εφαρμογής στο παρελθόν των κοινοτικών ταμείων. Θέλω να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπαν και οι δύο ε, βουλευτές και θα το πω στα πολωνικά για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Θα διευκρινίσω δηλαδή ποια είναι η άποψη της πολωνικής κυβέρνησης πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, η πολωνική κυβέρνηση, όπως λέει ο αναφέρον, θεώρησε ότι η προσβασιμότητα στην Ανατολική Πολωνία είναι πολύ σημαντική και για τη χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δομή των λειτουργικών προγραμμάτων όπως υποβλήθηκαν ειδικά για το λειτουργικό πρόγραμμα της Ανατολικής Πολωνίας όριζαν ότι σημαντικά κονδύλα θα διατεθούν για τα έργα υποδομών και επίσης θα υπάρχουν συγχρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής που θα καλύπτουν οδικά έργα. Υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος τέτοιων έργων που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν και έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κατάλογος. Άμα διαβάσετε αυτόν τον κατάλογο θα διαπιστώσετε ότι προβλέπονται χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής για τα σύνολα δίκτυα Ολοκλήρωσα το πρώτο λοιπόν σημείο μου, η πρώτη μου παρατήρηση. Άρα λοιπόν αυτός ο άξονας θα τύχει συγχρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και στα σύνολα δίκτυα και στα κομβικά. Δεύτερον, η συγχρηματοδότηση δεν εξαρτάται από το αν το έργο αυτό η εμπίπτει στα ολοκληρωμένα δίκτυα ή στα σύνολα δίκτυα ή στα κομβικά δίκτυα, στα επιμέρους δίκτυα. Είναι μέρος των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων, των TEN, όπως αποφασίσαμε για την, πενταετία, για την εξαετία 2007-2013 τότε αποφασίστηκε η συμπερίληψη στα τέν και συγχρηματοδότηση αυτού του έργου. Όσον αφορά λοιπόν το Connecting Europe Facility, είναι σαφές ότι αυτός ο φορέας, αυτό το μέσον μπορεί να χρηματοδοτήσει οδικά έργα. Δεν χρηματοδοτεί αποκλειστικά σιδηροδρομικά δίκτυα, αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Euro, Connecting Europe και οδικά έργα με τη βοήθεια επίσης του Ταμείου Συνοχής. Από όλες τις πολιτικές ομάδες της Πολωνίας είχε συμφωνηθεί ότι το Ταμείο Συνοχής θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση και η πολωνική κυβέρνηση επίσης. Θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση οδών στην Ανατολική Πολωνία και οδικών αξώνων όλες οι λεπτομέρειες του ποιοι δρόμοι και άξονες θα χρηματοδοτηθούν υπάρχουν και έχουν υποβληθεί. Έχουν ε, εγκριθεί, έχει εγκριθεί η συγχρηματοδότηση και πιστεύω ότι η ουσία αυτής της αναφοράς είναι αν θα πρέπει να καλυφθεί από το, το κομβικό ή το συνολικό δίκτυο. Αλλά για τη χρηματοδότηση έχουν ληφθεί αποφάσεις, δεν εμπίπτει στην αναφορά η πρόεδρος. Από ό,τι κατάλαβα εγώ υπάρχει μια πρόταση να κλείσει ο φάκελος. Έχω δύο, τρεις συναδέλφους να κλείσει ο φάκελος της αναφοράς και είναι η μόνη πρόταση που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Υπάρχει άλλη πρόταση παρακαλώ. Συμφωνείτε να κλείσουμε το φάκελο. Ο κύριος Πορέμπα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λυπάμαι κυρία πρόεδρε αλλά κατά την αρχική μου παρέμβαση είπα σαφέστατα ότι θέλω να παραμείνει ανοιχτός αυτός ο φάκελος. Άρα δεν είναι μόνο μία πρόταση να κλείσει ο φάκελος, υπάρχει και δική μου να μείνει ανοιχτός ο φάκελος. Συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, ναι ναι η παρέμβασή σας ήταν σαφέστατη και μακρά. Δύο προτάσεις λοιπόν έχω, η μία είναι να παραμείνει ανοιχτός ο φάκελος, η άλλη να κλείσει. Πιστεύω ότι το δίκαιο είναι να ψηφίσουμε. Και να σημειώσουμε ότι δεν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εδώ ε, είναι σωστά ε, τα, το δικαίωμα ψήφου. Όλες οι πολιτικές ομάδες. Το S&D έχει 9, το ΕΛΚ έχει τις σωστές ψήφους, 10 έχει το ΕΛΚ. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε με διανατάσεως χειρός ή αν θα κλείσουμε ή όχι την αναφορά. Παρακαλώ, ποιος, ποια μέλη μας θέλουν να κλείσει ο φάκελος. Ψηφίζουμε ποιο διανατάσεως χειρός να κλείσει ο φάκελος. δέκα. Και πόσοι από εσά θέλουν να μείνει ανοιχτό ο φάκελο τη αναφορά. Ένα, δι, δύο, τρεις. Αποχές, δύο. Τρεις. Μπορούμε να επαναλάβουμε, λέει η πρόεδρος. Αποχές, μόνο οι αποχές παρακαλώ. Νομίζω είδα τρία χέρια. Τρία. Ωραία, τρία. Εντάξει. Δέκα υπέρ του κλεισίματος. Α. μπορούμε ε, να ξαναψηφίσουμε, λέει ο κύριος Ποντέμα. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε, λέει η πρόεδρος. Και ρωτώ, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του κλεισίματος της αναφοράς. Το ΕΛΚ έχει 10 ψήφους. 10, όχι παραπάνω. Δέκα λοιπόν. Πόσοι ψηφίζετε να μείνει ανοιχτό ο φάκελος. Ένας. Όχι, τρεις. Αποχές παρακαλώ. Τρεις. Ωραία. Ε, το ίδιο αποτέλεσμα που είπαμε και πριν. Λοιπόν, η απόφαση παραμένει από της Επιτροπής Αναφορών να κλείσει ο φάκελος Υπερψήφισαν 10, καταψήφισαν 4, ε, αποχές 3. Α, καταψήφισαν 3, αποχές 3. Ένα λεπτό να φτιάξω εδώ το φάκελό μου για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Πού είναι, το 10. Για την Κύπρο Αμόχωστο. Αναφορά του Λοΐζου Αυξεντίου έξω ονόματος του κινήματος προσφύγων Αμοχώστου σχετικά με την απόδοση της κλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της. <clears throat> Δεδομένου ότι είναι απόν ο αναφέρον, μας έχει όμως υποβάλει γραπτό σε εμά, τη γραμματεία και σε μένα προσωπικά, ότι το θέμα αυτό θεωρείται εξαιρετικά επίγον ακόμα. Δεν είχε τον καιρό να έρθει εδώ και θέλει ο φάκελος να παραμείνει ανοιχτός. Για να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε όταν θα κινηθεί η υπόθεση η οποία είναι πολυδιάστατη Δεδομένου λοιπόν ότι είναι απόν ε, ο αναφέρον ε, θα αποτανθώ απευθεία στην Κομισιόν. Δεν έχω όνομα. Ποιος είναι από την Κομισιόν παρακαλώ παρόν. Η, κυρία Ντεμπούση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή έστειλε την απάντησή της το 2010, ήταν η τελευταία μας απάντηση σε σχέση με αυτή την ε, αναφορά και θα σας δώσω κάποιες ε, τελευταίες πληροφορίες. Το 2012 οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος υπό τον αιγίδα του ΟΗΕ ε, ανεστάλησαν στις 11 Φεβρουαρίου του το 2014 ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας συμφώνησε σε κοινόν εκκοινοθέν προκειμένου να επαναξεκινήσουν ε, πλήρες διαπραγματεύσεις. Οι δύο ηγέτες των κοινοτήτων έχουν επίσης ζητήσει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και συζήτησαν επίσης και το θέμα των βαροσίων. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σημειωθεί ακόμα κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ξεκίνησαν οι συζητήσει δεδομένη τη παρέμβαση τη Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου. Από το 2006 υπάρχει ένας κανονισμός του Συμβουλίου που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης περίπου 31 εκατομμυρίων ευρώ στο, ανάλογα με το ετήσιο δημοσιονομικό πλαίσιο και κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο έχει ε, διαχειριστεί αυτή την χρηματοδότηση προς τον τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να είναι ε, υποστηρίζει πλήρω τις προσπάθειες των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα ε, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η επιστροφή των σκληστής περιοχή της Αμοχώστου προς τους ε, κατοίκου τη είναι ένα από τα σημεία κλειδιά αυτή της διαπραγματεύση, Μια πλήρης λύση που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών θα ήταν ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος για να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένης και της ε, επιστροφής των βαροσίων. Η Επιτροπή έχει ασκήσει πιέσει και στους δύο ηγέτες των κοινοτήτων να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ξαναξεκινήσουν δομημένες ε, οργανωμένες διαπραγματεύσεις ώστε το δυνατό πιο γρήγορα έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε δίκαιη, πλήρη και βιώσιμη λύση του προβλήματος της Κύπρου. Υποστηρίζουμε πλήρως τις ενέργειες του ειδικού ε, εισηγητή, ανταποκριτή του ΟΗΕ, στην προσπάθειά του να γεφυρώσει τις ε, δύο κοινότητες της ρεπαγματεύσεις. Τον Φεβρουάριο η η Ευρωπαϊκή Ένωση στην δήλωσή της υποστήριξε την προσπάθεια να βρεθεί μια λύση με βάση τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια όθεση προς μια οριστική λύση που θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραμένει πάντα στη διάθεση ε, των κοινοτήτων έτσι ώστε να συνεισφέρει στην εξέβρεση τελικής και, πλήρους και συνολικής λύσης. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα κυρία Σακοράφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παράγραφο του σχέδιου συστάσης της Επιτροπής όπου λέει ότι εάν δεν υπάρξουν αυτά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή Αναφορών θα μπορούσε να επανεξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση και να μελετήσει τη δυνατότητα περαιτέρω ενεργειών, όπως παραδείγματος χάρη, να φέρει το ζήτημα των αναφερόντων της αμοχώς του στην Ολομέλεια. Κυρία Πρόεδρε, είναι περιττό να, να σας κουράσω με αναφορά στα όσα έχουν γίνει από τότε, τα οποία όμως θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά πάνω στο θέμα, ώστε να πούμε ότι συνιστούν πρόοδο. Δυστυχώς το Κυπριακό έχει καταντήσει παιχνίδι γεωπολιτικών και ενεργειακών συμφερόντων με τεράστια ευθύνη φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό. Θα περιοριστώ όμως να αναφερθώ στα της Επιτροπής και θα ε, επαναλάβω σημεία της αναφοράς. Σημειώνει η αναφορά ότι τα βαρόσια θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαστήριο ανάπτυξης και σύμβολο του μέλλοντος της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Προεδρία της, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστούν από κοινού στην κατεύθυνση αυτή. Και αυτού, αφού στη συνέχεια επισημαίνει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας με μνημόνευση των αλλεπάλληλων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καταλήγει με το συγκλονιστικότερο κατεμένα συμπέρασμα αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι και στις δύο πλευρές της νήσου οι άνθρωποι ξεχνούν πώς να συμβιώνουν και να μιλούν η μεν την γλώσσα των δε. Οι γενιές μεγαλώνουν σε ηλικία και πολλοί από όσου θυμόντουσαν την Κύπρο πριν από το 1974 έχουν ήδη πεθάνει. Επομένως, η κατάσταση είναι επίγουσα και κρίσιμη. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω και την Επιτροπή αλλά και τους συναδέλφους όλους στα πλαίσια των υποχρεώσεων και των δυνατοτήτων της Επιτροπής μας να συνταχθούμε και να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση των συμπερισμάτων της συγκεκριμένης της Επιτροπής μας δεδομένων των συγκυριών, των διεθνών συγκυριών, ε, δεν είμαι ούτε εθεροβάμων, αλλά ούτε και ρομαντική να πιστεύω ότι μπορούμε εμείς στην Επιτροπή μας να λύσουμε το θέμα της, του Κυπριακού, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά εάν συντονίσουμε τις ενέργειές μας και εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες των παρεμβάσεων που μπορεί να έχει η Επιτροπή μας, πιστεύω ότι ίσως μπορέσουμε, επιβάλλοντας μια δίκαια λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, να δώσουμε ένα δείγμα ανατολισμού στις περίπλοκες διαπραγματεύσεις που ελπίζω ότι πρέπει και θα ξαναρχίσουν. Δεν περιορίζουμε λοιπόν να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση, αυτό το θεωρώ αυτονόητο, αλλά να την δούμε σαν μια χρυσή ευκαιρία συμβολής από πλευράς μας στην ειρική διευθέτηση του ζητήματος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Κύριε Οργείο, ο λόγος είναι για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αυτό που θα πω σαν εισαγωγή δεν έχει να κάνει καθόλου με την εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά έχει να κάνει γενικά με την αναφορά όπως την άκουσα εκ μέρους της Κομισιόν. Ε, πραγματικά ε, χρειάζεται κανείς να έχει εκπαίδευση στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για να μπορέσει να καταφέρει να βγει έξω από το θέμα μιλώντας για το θέμα. Η αναφορά στις συνομιλίες δεν έχει καμιά σχέση με, το υποσυζήτηση, με την υποσυζήτηση αναφορά. Η αναφορά ζητά την επιστροφή των πολιτών μιας πόλης η οποία είναι περίκλειστη, ε, κατοικείται από φίδια και ποντίκια επί 40 χρόνια και θα πρέπει να επιστραφεί ανεξάρτητα από τη λύση του Κυπριακού. Θα πρέπει οι κάτοικοι αυτοί να δικαιούνται να πάνε στο σπίτι τους διότι αυτό δεν μπορεί να διασυνδέεται κατά ανάγκη με τη λύση του Κυπριακού, τουλάχιστον συζητώντας για την αναφορά. Ε, βρίσκω λοιπόν αδόκιμη την, την, την προσπάθεια να με το ζήτημα με μια συζήτηση ε, που έχει να κάνει γενικότερα με τις συνομιλίες, τις οποίες οπωσδήποτε και εμείς υποστηρίζουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι εν ώψη της ε, άποψης του αναφέροντος, όπως την μεταφέρατε εσείς εδώ, να παραμείνει το ζήτημα ανοιχτό, είναι και δική μας θέση, αλλά θέλω να υπομνήσω ότι στην προηγούμενη συνεδρία μας είχαμε συζητήσει για την ανάγκη ε, νέας επίσκεψης σαν fact-finding mission στην Αμόχωστο. Εμείς δεν και εγώ είμαστε, ούτε θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει αμάν-αμάν ή αύριο, αλλά μέσα στο 2015 να γίνει αυτή η επίσκεψη για να αναθερμανθεί αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό ζήτημα. Και θέλω να κλείσω για όσους συναδέλφους ίσως τώρα ακούν αυτή την υπόθεση ή δεν έχουν πολλές λεπτομέρειες. Ε, μιλάμε για μια πόλη ευρωπαϊκής ιστορίας που συνδέει αν θέλετε και την ιστορία της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή, με τη Συρία, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, με την Ελλάδα, με, την, ε, με τη Γαλλία τέτοιας, ιστορία, τέτοιας ιστορίας βάθος είναι η υπόθεση της του που πρέπει να το ξεμπλέξουμε από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα και να το δούμε σαν ανθρωπιστικό θέμα δικαιώματος των κατοίκων αυτής της πόλης να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, και πριν από τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ευχαριστώ. Κυρία Κυρικό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα μπορούσα να προσθέσω πολλά σε αυτά που είναι οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Απλώς να επισημάνω και εγώ ότι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρεται ρητά πως είναι ξεχωριστό ζήτημα η επιστροφή των κατοίκων της Αμοχώστου και στο ψήφισμα της δεκαετίας του 80 και στο ψήφισμα της δεκαετίας του 90, 84 και 92. Όπως επίσης και η δικιά μας ε, απόφαση της Επιτροπής ε, Αναφορών του 2008 που ανέφερε ακριβώς το ψήφισμα του 1984 σαν τη δυνατότητα των κατοίκων να επιστρέψουν ανεξάρτητα από τη λύση του Κυπριακού. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι πως η μη επιστροφή των κατοίκων δεν είναι μόνο η αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου για να βρουν μια κοινή βιώσιμη λύση που ελπίζουμε πως θα το καταφέρουν τελικά είναι η αποτυχία και του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο να μπορέσει να προωθήσει κάτι το οποίο σύμφωνα με τα ψηφίσματά του ήταν όριμο και ήταν σωστό να γίνει. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν συμφωνούμε και εμείς στο ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή ή να μείνει ανοιχτό το petition ακριβώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το Κοινοβούλιο από μόνο του θα αποφασίσει ότι το θέμα είναι κλειστό, ότι απέτυχε σε τέτοιο σημαντικό βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Mr. Το μέλλον της του είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Πιστεύω από τότε που επισκέφθηκαν την Κύπρο και συνελήφθη στα Βαρόσια όταν πέρασα ένα φράχτη για να δω να έχω η διαράψη από τον τουρκικό στρατό. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματο του συναδέλφου μα τη κυρία Θεοχάρου, η Ελένη Θεοχάρους, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα γιατί είναι στο Στρασβούργο και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματό τη. Αυτή η πόλη φάντασμα τη αμοχώ του βρίσκεται παράνομα υποκατοχή των τουρκικών στρατευμάτων που βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο από την εισβολή του 1974. Επομένως μόνο η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να λάβει αποφάσεις για το τι θα γίνει για αυτό το, σε αυτό το τμήμα της Κύπρου. Υπάρχει μια έκθεση την οποία έχει εκδώσει αυτή η Επιτροπή επί τη βάση της, επίσκεψης fact-finding που έγινε πρόσφατα, την προηγούμενη, η οποία όμως δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί οι τουρκικές αρχές δεν έδειξαν καμία διάθεση συνεργασίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η πρόταση Μία πρόταση λοιπόν που θα μπορούσα να σας κάνω κυρία Πρόεδρε για να συνεχίσουμε τη δράση μας σε αυτόν τον τομέα είναι να αποστείλουμε μια επιστολή στην τουρκική κυβέρνηση και να ζητήσουμε από την τουρκική κυβέρνηση γιατί δεν έχει λάβει κανένα μέτρο, έχει προβήσει καμία ενέργεια όσον αφορά το θέμα τη αμοχώς του και πιο συγκεκριμένα γιατί δεν έχει επιστραφεί η πόλη αυτή στους ε, νόμιμους κατοίκους της όπως ζητά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Τουρκία φέρει την νομική και πολιτική ευθύνη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Η δράση λοιπόν που προτείνουμε μπορεί να ανοίξει, πιστεύω, το δρόμο, να βοηθήσει στην εξέβρεση βιώσιμη ε, κοινή λύση του κυπριακού προβλήματος. Πιστεύω ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της Τουρκίας πριν να, τα επόμενα, πριν να προχωρήσουμε στα επόμενα μας βήματα. Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε ακόμα μια αποστολή διαρευνητική fact-finding γιατί δεν υπάρχουν νέα γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την αντίδραση των ε, τουρκικών αρχών και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους πιέσουμε με επιστολές, να ζητήσουμε εξηγήσει. Κατά βάση λοιπόν ζητώ κυρία Πρόεδρε να στείλουμε μια επιστολή στις τουρκικές αρχές ζητώντας τους εξηγήσει για την αδράνεια που έχουν δείξει στο θέμα αυτό. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος θα ήθελε τον λόγο. Παρακαλώ να καταλήξουμε λοιπόν στον συμπέρασμα ότι παραμένει ανοιχτή η αναφορά και ε, θα στείλουμε μία επιστολή προς την κυβέρνηση της Τουρκίας σύμφωνα και με αυτά που είπε ο κύριος Βαν Λέντσα θα αναφερθούμε επίσης και στα προτινόμενα συμπεράσματα από την προηγούμενη αποστολή που είχε γίνει επιτόπου εκεί, αναφορές δηλαδή στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταυτόχρονα εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας ζητήσω να προσθέσουμε εμείς από την Επιτροπή Αναφορών να στείλουμε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τι σκοπεύει να κάνει με την γραπτή δήλωση που έγινε εδώ και δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα βρούμε την ακριβή ημερομηνία και θα ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Ήταν μία από τις λίγες γραπτές δηλώσεις τις οποίες είχε αποδεχθεί επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτά. Ε, θέλετε κάτι άλλο. Θέλετε να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο είπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το EPRS, και δίνω το λόγο στον κύριο Ντάν. There you are, exactly. Hiding here, Chairman. Thank you. I'm happy Κρύβομαι εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εκτιμώ την κίνησή σας. Δεν θα κάνω μια πλήρη παρουσίαση. Θα ήθελα να σας δώσω λίγα, θα έλεγα κεφάλαια ε, για το τι κάνουμε. Εγώ αντιπροσωπεύω ένα νέο γενικό διευθυντή και μια υπηρεσία το EPRS, το οποίο βασίζεται στην αντίστοιχη ερευνητική υπηρεσία του Αμερικανικού Κογκρέσου, EPRS. Θα σας εξηγήσω γιατί. Εκπροσωπώ μια γενική διεύθυνση λοιπόν, μια διεύθυνση συγγνώμη, στο εσωτερικό της Γενικής Διευθύνσεως για τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Έτσι δημιουργηθήκαμε. Το τμήμα μας λέγεται Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία και Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Είναι απόφαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου του 2012. Έγινε μια ανάλυση τότε από το Προεδρείο και πολλοί συμφώνησαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια πολύ αποτελεσματική νομοθετική μηχανή με σωστό τρόπο ασχολείται με θέματα τροπολογιών, με θέματα συναποφάσεων, αλλά έχει ελλείψει σε επίπεδο ελέγχου ε, των αποφάσεων της εφαρμογής τους κτλ. Ο Γενικός Γραμματέας μας είχε κάνει μια πλήρη ανάλυση συγκρίνοντας ε, το τι γίνεται και στα υπόλοιπα κοινοβούλια και είπε ότι το Κογκρέσο ναι μεν έχει κάποιες δυσκολίες σε άλλους τομείς αλλά στον τομέα αυτό ήταν πρωτοπόρο. Εμείς λοιπόν θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια εμβριακή στην αρχή ε, υπηρεσία η οποία να μπορεί να δίδει στο Κοινοβούλιο περισσότερη προστιθέμενη αξία από ό,τι σήμερα. Το κάναμε με τρεις τρόπους καταρχάς. Υπάρχει η ενότητα European Added Value, Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία, που αξιολογεί τις ε, κοινοτικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες όπως η ε, οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας σύμφωνα με το 225 εμείς τους δίδουμε κάποιες μελέτες επιπτώσεων της πρότασης και εμεί τεκμηριώνουμε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να κατατεθεί στην Ολομέλεια. Έχουμε επίσης και τις λεγόμενες εξάντε μελέτες επιπτώσεων, εκ των προτέρων δηλαδή προληπτικών αν θέλετε, είναι ένα σύντομο σημείωμα, είναι 7-8 σελίδες και είναι κάτι το οποίο απλά συμπληρώνει την πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιολογούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραμμίζουμε ε, τα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν περισσότερης ε, προσοχής και μελέτης. Σημασία μεγαλύτερη έχει η λεγόμενη εκ των υστέρων αξιολόγηση, η ex post appraisal. Εκεί προσπαθούμε να δούμε το τι γίνεται με τις αποφάσεις αυτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι λέει για αυτές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συμφωνείται ότι έχει επίσημα, δεν έχει μάλλον νομοθετικές αρμοδιότητες, αλλά στην ουσία είναι σε θέση να να πάρει αποφάσεις νομοθετικής φύσεως σαν Συμβούλιο. Δεύτερον έχουμε επίσης και μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε επίπεδο ελέγχου των επιπτώσεων των αποφάσεων τις οποίες έχουμε λάβει και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τροπολόγησης ή αναθεώρησης των νομοθετικών ρυθμίσεων παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους έχουν γίνει οι αλλαγές αυτές. Και τέλος και βασική μας αρμοδιότητα εδώ είναι η ίδια η εφαρμογή των νομοθετικών αποφάσεων, η εκ των υστέρων δηλαδή ε, έρευνα. Είναι κάτι το οποίο συμπληρώνει τις εκθέσεις εφαρμογής που πολλές φορές υπάρχουν σε ορισμένες επίτροπες. Στο παρελθόν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες εκθέσεις μία φορά το χρόνο, τώρα δεν υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των εκθέσεων εφαρμογής τις οποίες μπορούν να συντάξουν οι, Ευρωπα... οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεργαστούμε και με τη δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή. Εσείς είσαστε πραγματικά το πρόσωπο της ε, Ένωσης απέναντι στους πολίτες που αποδεικνύει στους πολίτες το πώς τους επηρεάζουν οι κοινοτικέ νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος της EPRS είναι να βοηθήσει λοιπόν τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Προς το παρόν λειτουργούμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως είπα έχουμε περιορισμένους πόρους αλλά έχουμε αρχίσει να αυξάνουμε τις, ε, τον αριθμό των ε, μελετών μας σε σχέση με τις μελέτες επιπτώσεων και τις αξιολογήσεις τα τελευταία δύο χρόνια και νομίζω ότι η ενασχόλησή μας και με τα θέματα εφαρμογής είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει θετικά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, σύντομα ήταν αυτά. Εμείς ήρθαμε εδώ βασικά για να ακούσουμε τις προτάσεις σας, τις εκτιμήσεις σας και ίσως και τις συμβουλές σας. Εδώ έχω τον ε, κύριο Όμπριχτ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των πολιτικών και ε, παρακαθήμενος είναι ο αρμόδιος για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Λοιπόν, ελπίζω να ήμουν κατανοητός πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μία τελευταία λέξη ε, στην είσοδο μπαίνοντας θα δείτε ε, ένα εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει ακριβώς τις ε, δραστηριότητές μας για διάφορα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και σίγουρα και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι αναμένετε μπορεί να έρθουμε να σας ζητήσουμε τη βοήθειά σας, τη συμβουλή σας. Προσλέπω λοιπόν με μεγάλη χαρά στην περαιτέρω συνεργασία και δίνω το λόγο στον κύριο Βαλέντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως, θα είμαι τηλεγραφικός. Έχουμε ένα θαυμάσιο μέσο στη διάθεσή μας, αυτό το κέντρο, το υπηρεσία ερευνών, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για θέματα που είναι σημαντικά και πιστεύω όλοι να ακούσαμε με προσοχή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εργαλείο που είναι στη διάθεσή μας, αυτή την υπηρεσία. Η Πρόεδρος, είναι θαυμάσιο πράγμα να ε, τελειώνει η συνεδρίαση με θετικό τόνο, με μια θετική ατμόσφαιρα πριν από χρόνια εργαζόμουν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ήμουν μέλος στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και πάντοτε μου άρεσαν αυτά τα ε, θέματα τα οποία έχουν μια θετική εξέλιξη και τώρα ειδού άλλη μια ευκαιρία συνεργασίας. Ε, περιέργως είμαστε ε, τελειώνουμε νωρίς σήμερα. πώ έγινε αυτό δεν ξέρω, αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την βραχνάδα μου, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι καλύτερα αύριο. Α ξεκουραστούμε όλοι λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλό σα βράδυ.